Voilà. Alors l'ordre du jour τη ημερήσια διάταξη θα προχωρήσουμε τώρα σε, στη δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή και είπα τη εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Ο κ. Πίμπαλκ στην αντικαθιστά τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Κύριε Επίτροπε, σα δίνω το λόγο για να μιλήσετε εξ ονόματο τη Αντιπροέδρου. Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Η εξαετής ε, μεταβατική περίοδος μετά τη συμφωνία στο Σουδάν ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το Σουδάν αλλά και για την Αφρικανική Ήπειρο συνολικά. Ο λαός του Νοτιού Σουδάν περίμεναν πολλά χρόνια τη στιγμή αυτή. Η ανεξαρτησία της χώρας θα ανακηρυχθεί στις 9 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιπροσωπεύεται στην ε, τελετή της ανεξαρτησίας από την ύπατη εκπρόσωπο και την πρόεδρο της Επιτροπής. Μετά από ένα αξιόπιστο δημοψήφισμα στο ξεκίνημα του έθνους, συγχαρήκαμε τα δύο μέρη για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν στη διοργάνωση του δημοψηφίσματος. Καλωσορίζουμε το ότι ο πρόεδρος Μπασίρ δημόσια δήλωσε ότι το Βόρειο Σουδάν θα είναι η πρώτη χώρα που θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Νοτίου. Ωστόσο, αμέσως μετά το δημοψήφισμα η θετική άβρα εξαφανίστηκε. Υπάρχουν ανησυχητικές τάσεις εντάσεων και συγκρούσεων. Οι πρόσφατες συγκρούσεις στον στο ΑΕΡΑΜ και, την αμπίγια μπορεί να οδηγήσουν σε νέες συγκρούσεις μεταξύ Βορρά και Νότου. Συζητήσαμε το Σουδάν στο Συμβούλιο Εξωτερικών και τον Ιανουάριο και τον Μάιο θα επανέλθει το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών ε, της 20 Ιουνίου. στο, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο θα παρουσιάσει τότε μια συνολική προσέγγιση στρατηγική τη Ένωση για το Σουδάν με έμβαση κυρίω στο ανεξάρτητο Νότιο Σουδάν, αλλά περιλαμβάνοντα και στοιχεία επικοδομητική εμπλοκή μα και στο Βόρειο Σουδάν μεταξύ και και των μεταβατικών καταστάσεων στο Νταρφούρ και στην Ανατολή. Θα έχουμε δηλαδή μια συνεργασία δύο σε, και με τα δύο κράτη. Η προσέγγιση αυτή θα είναι ένα στρατηγικό κείμενο που θα περιλαμβάνει τα βασικά ε, θέματα της πολιτικής μας προς, το Σουδάν, προς τα Σουδάν. Στο στόχος θα είναι η ειρήνη μεταξύ των δύο κρατών και ο εκδημοκρατισμός και η ευημερία και στις δύο χώρες. Θέλουμε να υπάρχουν, να συνυπάρχουν ως καλοί γείτονες δύο ειρηνικά κράτη με ανοιχτά σύνορα που επιτρέπουν τις διασυνοριακές ανταλλαγές ατόμων, αγαθών, κεφαλαίου και ιδεών. Το Νότιο Σουδάν θα χρειαστεί την προσοχή μας για να σταθεροποιηθεί, να βελτιωθεί η θεσμική ε, λειτουργικότητά του και να μην έχουμε ένα νέο ε, διαλυμένο κράτος. Η στρατηγική μας θα είναι να εξετάσουμε μια σειρά σημαντικών στοιχείων. Η ενίσχυση της παρουσίας της Ένωσης στην Τζούμπα με την σύσταση αντιπροσωπείας της Ένωσης. Να ξεκινήσουμε έναν ολοκληρωμένο πολιτικό διάλογο με συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία ε, και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για τη σταθερότητα της περιοχής αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Διαθέσαμε συνολικά ε, επιπρόσθετα 200 εκατομμύρια ευρώ για τον Νότιο Σουδάν. Αθρηστικά δηλαδή 300 εκατομμύρια στο σύνολο. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη σε ένα κοινό πρόγραμμα για την μεγιστοποίηση του αντικτύπου της βοήθειας αυτής. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και θεωρούμε ότι το εμπόριο πρέπει να είναι κομμάτι της προσέγγισης αυτής. Προφανώς θα υπάρξουν απώλειες για το Βόρειο Σουδάν. Πρέπει ωστόσο να βοηθήσουμε τους μεταρρυθμιστές στο Βορρά, να προωθήσουμε έναν γενικό πολιτικό διάλογο και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση του Χαρτούμ. Η πρόσφατη επίσκεψή μου ήταν και ένα μήνυμα εμπλοκής τη Ένωση μετά τη θετική ανταπόκριση του Χαρτούμ στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Μα ανησυχεί η βία, η πρόσφατη βία και οι συγκρούσεις που αποτελούν παραβίαση της Συμφωνίας Ειρήνης. Ζητούμε από τις δύο πλευρές να μην προχωρήσουν σε άλλες προκλήσεις και να διαπραγματευτούν μακροχρόνια την συνύπαρξη την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων που ζουν κοντά στην Αμπίγια και μέσα στην Αμπίγια. Σε ό,τι αφορά την κράτηση δημοσιογράφων ή υπερασπιστών των δικαιωμάτων του, του ανθρώπου, θεωρούμε ότι βασική αρχή της συμφωνίας είναι η δημιουργία δημοκρατικής κυβέρνησης που θα στηρίζεται στις βασικές ελευθερίες. Θέλουμε να υπάρξει θεσεβασμός των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και της, ε, του εκδημοκρατισμού και στο Βόλιο και στο Νότιο Σουδάν. Επίσης, να αναφερθώ στον Ταρφούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη βία στον Ταρφούρ που οδηγεί σε μετατοπίσεις πληθυσμού και στην ε, ανθρωπιστική κρίση. Τα καλά νέα είναι ότι τρεις Ευρωπαίοι πολίτες που ήταν όμοιροι στον Ταρφούρ τους τελευταίους μήνες απελευθερώθηκαν. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στον Ταρφούρ, εξασφαλίζοντας θετικά, θετική έβραση της ειρηνευτικής διαδικασίας και επιτρέποντας να υπάρξει εξέλιξη των πολιτικών συζητήσεων επιτόπου. Θέλουμε στην διάσκεψη των δωρητών να υπάρξει λύση και να υπάρξουν εξελίξεις για μια, εξελίξεις για μια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Να, να αναφερθώ στο θέμα της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να επιτευχθεί η μόνιμη ειρήνη στον τροφού χωρίς δικαιοσύνη και ε, συμφιλίωση. Πρέπει να υπάρξει, να τεθεί τέρμα στην ατιμορρησία και ζητήσαμε να εμπλακεί η κυβέρνηση του Σουδάν στην, να συμμετάσχει πλέον στην καταδίωξη και σύλληψη των εγκληματιών πολέμου βάσει του ψηφίσματος 1503 του ΟΗΕ. Η βιώσιμη ειρήνη και η δικαιοσύνη είναι βασικές προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, στο... λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία θα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτρο αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν ο η χαρά, ο ενθουσιασμό των πληθυσμών. Ήταν ευτυχεί οι άνθρωποι γιατί για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Μετά από 20 χρόνια πολέμου, για πρώτη φορά είχαν εντύπωση ότι αυτό που έλεγαν θα εισαγωστεί. Αυτά τα εκατομμύρια των Νοτιοσουτανών ε, δεν πρέπει να του απογοητεύσουμε. Δεν πρέπει όμω να ξεχνάμε χάσουμε και τους κατοίκους του Βορρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διαπραγματεύσεις να είναι κατά για να υπάρχει μια σταθερή βάση για τη μελλοντική εξέλιξη και σε κάθε μία από τις δύο νέες χώρες στη σχέση μεταξύ τους και στη σχέση της διεθνούς κοινωνίας και με τις δύο αυτές χώρες. Η βιωσιμότητα και η σταθερότητα του Βορρά και του Νότου είναι πρωταρχική σημασία. Είναι σημαντικό τα θέματα που δεν έχουν επιληθεί μέχρι στιγμή να επιληθούν. Το θέμα της υπηκότητα, του κατευθυνσμού του χρέου και των εισόδων του πετρελαίου ή και το πρόβλημα με τι μη καθορισμένα σύνορα. Από την άλλη μεριά, τα διαποσμήματα που θα γίνουν στο ΒΕΙ και το θα πρέπει να γίνουν. Η ε, κατάσταση της ΑΒΕ είναι πάρα πολύ ενισχυτική. Επιδεινώνεται από μέρα σε μέρα και πρέπει να περιμένουμε το σημείο χωρίς επιστροφή οι εντάσεις αν γίνουν ανοιχτή διαμάχη θα απειλήσουν την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν και να ξαναθέσουν τη χώρα σε χάος. Αλλά δεν πρέπει να συγκεντρώνουμε προσοχή μας μόνο στο ΑΠΙΑΙ και να μην ξεχνάμε τι γίνεται στο Νταρφούρ. Όπως είπατε και εσείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα προώθησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού διαφανείς διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ των δύο χωρών, η πάυση των, της βίας και καλή συνεργασία μεταξύ των δύο ετών είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση ώστε οι δύο αυτές χώρες να μπορούν πραγματικά να μετατραπούν σε πραγματικές χώρες μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας του πολιτικού πλουρισμού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Δεκάζαρ. Τρία λεπτά. Le 9 sud du Soudan célébrera θα γιορτάσει ξανά λοιπόν την ανεξαρτησία του το Νότιο Σουδάν και ανακτά την αξιοπρέπειά του. Κύριε Πίμπαλσκ, είχα προετοιμάσει μία ανακοίνωση τριών λεπτών, αλλά όταν σας άκουσα αναρωτιόμουν αν έπρεπε να πω κάτι. Θέλω να σας συγχαρώ γιατί ομολογώ ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον τρόπο τον οποίο ρυθμίστηκε το θέμα του Σουδάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω μαζί με τον λαό του Σουδάν να τον οδηγήσουμε στην ανεξαρτησία. Αναφερθήκατε στα βασικά προβλήματα, στο πρόβλημα της IBA που δεν έχει επιληθεί και στις πολιτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν για θέματα της ιδιότητας του πολίτη, του χρέους κτλ. Αναφερθήκατε επίσης και σε αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε στον αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό τομέα. Μιλήσατε για τη δικαιοσύνη, είπατε επίσης ότι δεν θα πουλήσουμε ε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ε, την ουσία την είπατε κύριε Πίμπαλξ. Για το θέμα της ανάπτυξης και για το θέμα το ανθρωπιστικό είναι αλήθεια ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν στο Νότιο Σουδάν και θα πρέπει να μην ξεχνάμε και να μην απομονώσουμε τον Βορρά. Όλα θα πρέπει να γίνουν γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, περιοχές που έχουν πετρέλαιο, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν δρόμοι. Οι προσδοκίες του πληθυσμού είναι τεράστιες και δεν θα πρέπει να διαψευστεί και να απογοητευτεί ο πληθυσμός αυτός από την ανεξαρτησία. Η ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι βασική μας προτεραιότητα και θα παραμείνει για πολύ καιρό για τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων των γυναικών, ε, του πολιτικού πλουραλισμού. Ξέρετε ότι στο Νότο υπάρχει πολυγαμία. Οι γυναίκες αγοράζονται με ανταλλαγή αγελάδων. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν τα οποία θα πρέπει να μείνουν ε, δεν μιλάμε μόνο για την άμεση πολιτική δραστηριότητα, πολλά θα πρέπει να αλλάξουν. Όλα αυτά είναι δύσκολο να αλλάξουν, αλλά είναι ταυτόχρονα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Εγώ συναντήθηκα με την εκλογική επιτροπή του Νότου και του Βορρά βέβαια, αλλά κυρίως του Νότου. Θέλουν να νομοθετήσουν, θέλουν να έχουν ένα καλό σύνταγμα, θέλουν να χτίσουν τη χώρα τους και μας λένε ότι θα έχουμε αρκετά χρήματα, αλλά παρόλα αυτά βοηθήστε μας όντας μαζί μας. Και εσείς μέχρι τώρα έχετε αποδείξει ότι θα βοηθήσετε. Πήγατε εκεί, πήγε και η κυρία Γεωργίευα στο παρελθόν, θα πάει και η κυρία Άστον στην επέτειο της ανεξαρτησίας, στην εορτή της ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι η στρατηγική την οποία παρουσιάσατε για τον Νότιο Σουδάν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Θέλουμε μια παρουσία συνεχή, δεν θέλουμε μια, ένα ενσταντανέ της κατάστασης και μια στιγμιαία παρουσία τότε μόνο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί αυτά τα οποία κάνατε πολύ καλά είναι και είμαστε υπερήφανοι για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστώ κύριε Αντεκεζέρ. Ο κύριος Βάιλ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στις 9 Ιουλίου θα κλείσει ένα κεφάλαιο ακόμα της απικιακής διαδοχής. Μετά το δημοκρατικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το Νότιο Σουδάν να ανοίξει μια σειρά θεμάτων και να συζητήσει με το Βορρά χωρίς συγκρούσεις και να αποφευχθούν οι μεταναστευτικές κινήσεις. Το πετρέλαιο μπορεί να βοηθήσει και το βορρά και το νότο, φτωχές χώρες και τις δύο. Η Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουν τις χώρες να ενισχύσουν την, ε, τον πλουραλισμό και τις, τους δημοκρατικούς θεσμούς. Μια μεγάλη πρόκληση όταν η περιοχή ευρύτερα αντιμετωπίζει νέα προβλήματα. Βρισκόμαστε σε μία καθοριστική στιγμή. Δεν έχει λυθεί, δεν έχουν λυθεί τα ζητήματα. Συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος, ουσιαστικός κίνδυνος συγκρούσεων. Το Σουδάν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Πρέπει να παραταθεί η εντολή της αποστολής του ΟΗΕ. Οι κυβερνήσεις και στο Χατούμ και στη Τζούμπα πρέπει να δεχθούν τώρα την ε, παρουσία του ΟΙΕ, ο κύριος Ντέβα, ένα λεπτό. Σωστά τα λέει ο κύριος Πίμπαλκ. Είναι η... Έχουμε μπροστά μας μία από τις βασικές προκλήσεις της Ένωσης. Ως εισηγητής στο Κοινοβούλιο, πιστεύω για την εθνοδημιουργία, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για μας να βοηθήσουμε την δημιουργία του κράτους του Νότιου Σουδάν και να μετατρέψουμε τη συζητήση σε πραγματικότητα. Πρόκειται για μια χώρα πλούσια σε πρώτες ύλε, αλλά και με εξαιρετικά κακούς κοινωνικούς δείκτες. Ένα παιδί που γεννιέται εκεί σήμερα έχει περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει πριν το σχολείο παρά να φτάσει στο δημοτικό. πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολιτική ε, αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή στην αγορά πουλούνται ε, τρόφιμα που προέρχονται από την επιστημιστική βοήθεια. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ε, ενίσχυση όλων των δομών που χρειάζεται ένα νέο κράτος. Κράτος δικαίου, διαφάνεια, ε, εμπειρογνωμοσύνη. Ως εταίροι πρέπει να μας καλέσουν και να τους δώσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ήμασταν, ε, είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε ε, όταν μια χώρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Το θέμα εδώ βέβαια είναι ότι το Νότιο Σουδάν έχει στις πλάτες του μια πολύ βαριά κληρονομιά και φοβάμαι ότι η γιορτή την οποία θα θέλαμε να κάνουμε ίσως να μην αρμόζει λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή. Το Σουδάν, το Βόρειο Σουδάν αν θέλετε, επετέθη στην περιοχή του Αϊμπέη, το Νότιο Σουδάν αντέδρασε και το θέμα είναι να δούμε πόσο θα κρατήσει η κατάσταση αυτή. Η διεθνής κοινότητα έλεγξε τον τρόπο με τον οποίο ε, διαξήχθη το δημοψήφισμα, αλλά το θέμα του eBay δεν πήρε απάντηση και αυτό φοβάμαι ότι θα είναι πηγή πολλών μελλοντικών συγκρούσεων οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να μεταβούν επιτόπου για να ηρεμήσουν την κατάσταση και η απόφαση ελήφθη και αυτό είναι κάτι το θετικό. Αλλά θα πρέπει να μην παραγνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος. Το Σουδάν ε, θέλει να επηρεάσει με άμεσο τρόπο το μελλοντικό δημοψήφισμα στο fast als je dat Υπάρχει, ένα θέμα με κάποια κατηγορία του πληθυσμού που κατοικεί στην περιοχή του Αϊμπάι ε, και πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση εκεί ετείνει στο να περιπλακεί ακόμα περισσότερο θα πρέπει να υπάρξει επίσης διαγραφή του χρέους πάρα πολύ απλά για τον Νότιο Σουδάν. Το χρέος το οποίο στην ουσία συνήφθη από, την, από το καθεστώς του Χαρτούμ και το οποίο δεν εξυπηρέτησε φυσικά τους γεωργούς του Νότου. Και ένα τρίτο θέμα είναι το τι θα κάνουμε με τον πλούτο ο οποίος βρίσκεται στο, στο Νότιο Σουδάν, στο υπέδαφος του Νότιο Σουδάν. Ε, μπορούμε ας πούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες ε, του πρωτοκόλου διαφάνειας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις εξορρυκτικές δραστηριότητες και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια προς το βόρειο αλλά και το νότιο, στο νότιο αλλά και στο βόρειο Σουδάν να οδηγήσει σε τίμιες εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή αυτή. Πρόεδρε, νομίζω ότι ε, βλέπουμε τα πράγματα στην περιοχή αυτή με κάποιο φόβο πλέον μετά από τον αρχικό ενθουσιασμό. Ελπίζω όμως κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ξαναγιορτάσουμε. Ευχαριστώ κυρία Σαρζεντίνη. Κυρία Τσίμερ, ένα μισή λεπτό. Όλοι με μεγάλη ανησυχία ατενίζουμε αυτή την περιοχή του κόσμου και ξέρουμε ότι ο κίνδυνο ενό εμφυλίου πολέμου δεν έχει ακόμα αποφευχθεί. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ευάλωτη η ειρηνευτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει, όπω καταδεικνύουν και τα γεγονότα του Αμπιέη. Η διαμάχη εκεί είναι δραματική. Ο στρατό του Νοτιού Σουδάν έχει καταλάβει το Αμπιέη και υπάρχουν 50.000 ανθρώπων που είναι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να φροντίσουμε η πιστιστική και ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες να ξεκινήσει το γλωγορότερο δυνατόν. Και η έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες θα πρέπει να χορηγηθεί αμέσως. Ε, ήδη χωρί αυτές τις εντάσεις, το 40% του πληθυσμού του Νοτιού Σουδάν εξαρτάται από την επιστημική βοήθεια. Και το Νότιο Σουδάν θα είναι μια από τις πιο φτωχέ περιοχέ και χώρε του κόσμου και αν θέλουμε να παρέμβουμε είναι απαραίτητο η πόροι που διαθέτει το Συμβούλιο, τα 200 εκατομμύρια αυτά, για την επιστική ασφάλεια, για την παιδεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της χώρας να δαπανηθούν πραγματικά για αυτούς τους στόχους. Εμείς ως πολιτική ομάδα ζητούμε την άμεση απόσυρη των ε, ενόπλων δυνάμεων και του Βορρά και του Νότου από το ΑΠΤΖΕΙ. Και εν ε, Ενδεχόμενη παράταση τη εντολή του ΟΗΕ, του Ηνωμένων Εθνών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλοι οι παράγοντες αυτοίς που αφορούν το Κονγκό. Επίση, ένα σχετικό είναι ότι στο ψήφισμα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία έντονη απέτηση για τη διαγραφή του χρέους και για την εξέταση του εξωτερικού χρέους. Αυτό μου φαίνεται λυπηρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ. Το λόγο του Μπέλτερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν η σημερινή κατάσταση στο Σουδάν. Πρώτο ερώτημα. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Σουδενική κυβέρνηση την απελευθέρωση ενός ατόμου που ε, συνελήφθη σε ένα στρατόπεδο προσφύγων της 15 Απριλίου ε, κάποιος που συνελήφθη εκεί βασανίστηκε και έχει μεταφερθεί στο Καρτούμ. Οι γνώστες κατάσταση στο Νότιο Σουδάν είπαν ότι στην διαμάχη αυτή στο Αβιγέι ε, έχει ε, ε, διπλωματική πίεση προς τον κυβέρνηση του Αλπαζίρ, η οποία πίεση όμως δεν είναι καλά συντονισμένη. Έτσι λένε οι γνώστες της κατάστασης. Ε, φαίνεται ότι ο κύριος Μπασίρ θέλει την εντύπωση ότι δεν θα κάνουμε τίποτα κατά αυτού ή θα πρέπει να αυξήσουμε την διεθνή πίεση κατά του κύριο Μπασίρ. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Πρώτα σε ευχαριστώ. Οι, οι άλλοι μιλικές τώρα. Ο κ. Μάουρο πρώτα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να σημειώσω την ρεαλιστική προσέγγιση στην παρέμβασή σας και να κάνω δύο προτάσεις για να αξιοποιήσουμε και το λαμπρό έργο της συναδελφού κ. Δεκάιζερ τον τελευταίο καιρό έργο παρακολούθησης ε, του, της εμπειρίας του δημοψηφίσματος που ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για μένα τουλάχιστον και για το θεσμικό όργανο του Κοινοβουλίου. Δεν ξεπλάγει από το ότι μετά το δημοψήφισμα είχαμε μια μεταγενέστερη φάση ε, εντάσεων από πλευράς των ε, Σουδανικών αρχών, κυρίως στην Αμπιέγε ένα τμήμα της πολιτικής του χαρτούν είναι πάντα το stop and go. Πρώτα να δίνεις κάτι, μετά να, να, ένα στυλ που οδήγησε στην καταστροφή στο Νότιο Σουδάν. Προτείνω ωστόσο. Στην υπηρεσία εξωτερική δράση δημιουργήσαμε μια δομή που ασχολείται ρητά με την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων. Η δομή αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει τώρα στο BA, όχι όταν έχουμε μια πραγματική καταστροφή. Να υπα... ε, ξεκίνησε, λειτουργεί σωστά, είδαμε τι έγινε, πώς αντιμετώπισε την κρίση στη Λιβύη. Θα πρέπει η δομή αυτή να μπορεί σήμερα να ετοιμάσει ένα σχέδιο και να το παρουσιάσει στην Επιτροπή Εξωτερικών, εξεγώντας τι πρέπει να κάνει και δίνοντας τι δείχνοντας τι αξία μπορεί να έχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης όταν θέλουμε όλοι να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Μια άλλη τελευταία ε, σύσταση. σχέσεις μας με την Κίνα. Παντού λένε ότι η Κίνα έχει μεγάλο ρόλο στο Σουδάν και το λένε αυτό σαν να είναι ένα φάσμα που πρέπει να φοβόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πολύ προνομιούχες και, και καλές σχέσεις με την Κίνα, διότι πέραν των οικονομικών συμφερόντων θα πρέπει να θέσουμε και το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κύριε Γκόμες, 1,5 λεπτό. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Σουδανική κυβέρνηση, να αποσύρει τα στρατεύματα από το Αμπίγε. Η λύση στο Αμπίγε είναι αναγκαίο για να μην υπάρξει κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών και θέτοντα έτσι σε κίνδυνο τη διαδικασία που ξεκίνησε με το δημοψήφισμα. Οι πυροβολισμοί κατά του ελικοπτέρου του ΟΗΕ τον Μάιο είναι απαράδεκτη και πράξη δηλού. Είναι απαράδεκτη όπως είναι απαράδεκτη και το αίτημα των αρχών του Χαρτούμ να, φύγουν, να φύγει η παρουσία του ΟΗΕ από την περιοχή. Εκεί χρειάζεται ο ΟΗΕ περισσότερο από ποτέ για να παρακολουθεί την εξέλιξη και να εμποδίζει την επέκταση των συγκρούσεων. Η εξασφάλιση ειρηνικής μετάβαση στην εξαρτησία στο Νότιο Σουδάν απαιτεί επίσης να συνεχίσουμε να βάζουμε μπροστά στην ημερήσια διάταξη την μάχη κατά της ατιμορρησίας και για τις δύο χώρες και η Ένωση δεν θα πρέπει να κάνει καμία συμφωνία συναλλαγής με τον πρόεδρο Μπασίρ ε, για το οποίο θα περιλαμβάνει ότι, το ότι θα γνωρίσουμε την ανάγκη παραπομπής του ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για με τις κατηγορίες των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας του Νταρφούρ κατά του Σουδανικού λαού. Ο κύριος Γκέρενς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόσφατο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Σουδάν εγκαινιάζει μια νέα περίοδο θα έλεγα, ένα νέο στάδιο κάτι το οποίο το εσωτερική υπόθεση του Σοδάν με τη δημιουργία ενός νέου κράτους γίνεται αυτόματα διεθνής υπόθεση. Κάθε σχέση στον τομέα της ασφάλειας με το Χαρτούμ είναι κάτι το οποίο αφορά το διεθνές δίκαιο πλέον. Χαιρετίζουμε λοιπόν τον τρόπο που οι διάφοροι ε, εταίροι της διεθνούς κοινότητας ε, έχουν αφοσιωθεί στην προσπάθεια αυτή πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το νέο κράτος. Καταρχάς, η διαιτησία του κυρίου Μπέκη, Προέδρου της Νοτιού Αφρικής και εκπροσώπου της Ένωσης για την Αφρική Ενότητα, όπως επίσης και της κυρίας Ρόζα Λιπάτσεν που είναι η ε, ειδική εκπρόσωπό μας στο Σουδάν. Δεύτερον, η συμμετοχή του νέου κράτους στη Συμφωνία του Κοτονού δίνει νέες δυνατότητες συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να επικυρώσουμε άμεσα τη νέα αυτή προοπτική. Τρίτον, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικής ικανότητας των τεράστιων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η νέα χώρα ή τόσο εύθραυστη. Εδώ η τοσο εθραυστη εδω κοινότητα θα πρέπει να παρέμβει. Τέταρτον, Υπάρχει ανάγκη να παρέμβουμε και στην ανάπτυξη του Βορρά. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το Βορρά, ο οποίος αυτή τη στιγμή συντάσσει ένα νέο σύνταγμα. Η κατάσταση δραματική στον τομέα της ασφάλειας, στον Ταρφούρ, και η μονομερής κίνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ένα δημοψήφισμα στις αρχές Ιουλίου του 2011. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω τον σημαντικό ρόλο του Επιτρόπου, του Αρμοδίου, που ε, θεώρησε ότι αυτή η τόσο αποφασιστική περίοδος για το Σουδάν είναι και περίοδος δοκιμασίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βαντάλεν, ένα λεπτό. Ε, φτάνουμε στις 9 Ιουλίου, θα γίνει επίσημα ανεξάρτητο το Νότιο Σουδάν, θα γίνει μια χώρα ε, χριστιανική μια χώρα όμως η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Η παλιά αλεπού της πολιτικής στην περιοχή, ο Ομάρ Μπασίρ, δεν θα αφήσει να του ξεφύγει η ευκολιλία. Ήδη προσπάθησε να διώξει κόσμο από την περιοχή του Αϊμπέη, έχει ξεκινήσει μια εθνοκάθαρση στην περιοχή για την φυλή των Νίνκα και η ζωή στην περιοχή είναι πλέον ανασφαλής. Η κυρία Αστόν ξέρει ότι υπερασπιζόμεθα την πολιτική της για την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πέρα από αυτά τα οποία έγιναν στην Μπενγάζη πρέπει να κάνει συγκεκριμένες επιλογές και εις βάρος του ο Μαρμπασίρ γιατί ο λαός του Νοτίου Σουδάν πρέπει να υποστηριχθεί όσο καλύτερα γίνεται. Η κυρία Λόζινγκ, ένα λεπτό. το Φεβρουάριο πολλοί και εδώ στο σώμα ήταν πλήρες ελπίδων αλλά και ανησυχίες για το μέλλον του Σουδάν. Ο κίνδυνος βιαίων διαμαχών εκτιμήθηκε διαφορετικό. Είναι σαφές όμως ότι οι πολίτες του Σουδάν βρίσκονται ενώπιον προβλημάτων και χρειάζονται υποστηριχή μας. Τώρα τους βλέπουμε πάλι στις πρώτα σέλιδα των εφημερίδων γιατί έχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν με όπλα. Χαιρετίζω γι' αυτό την πρόσφατη ε, συμφωνία που επιτευχθεί με την ε, διατησία της ε, Νοτιοαφρικανικής Ένωσης μεταξύ Νοτιού και Βορείου Σουδάν. γιατί ακόμα και μια δύναμη Σμουνίκ των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί παρά να βλάψει όπως είδαμε στο Κονγκό. Θα πρέπει τα συμφέροντα των πολιτών του Βορρά και του Νότου να είναι στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας και όσον αφορά τις ε, ουσιαστικές ε, και όσον αφορά τις διπλωματικές ε, προσπάθειες. Ζητούμε την κατάπαυση της συνεργασίας μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Ευχαριστώ κύριε Λέζον. Πρόεδρο, κύριε Στρίφλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν μπορούμε παρά να χαρούμε για την ε, ειρηνική και αξιόπιστη ε, ε, οργάνωση του δημοψηφίσματος Τώρα υπάρχουν βέβαια προβλήματα όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση του νέου χώρου, της νέας χώρας και τις σχέσεις ε, της ε, χώρας αυτής με τους γειτονές σας και την κατάσταση στο ΑΠΕΗ που έχει πάρα πολύ πετρέλαιο. Οι κύριες ε, προκλήσεις είναι η ασφάλεια και ο σεβασμός των ανθρωπιστικών ερχών. Η κρίση δεν έχει αποφευχθεί. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να, εξασκεί, να ασκεί πίεση και να βοηθά ανθρωπιστικά κάτω των δυνατών. Η κατάσταση είναι δραματική, αλλά θα μπορούσε να επιδεινωθεί και να απειλήσει τη σταθερότητα τη περιοχή. Επίση, είναι σημαντικό η αναπτυξιακή βοήθεια που θα δοθεί στο Νότιο Σουδάν να είναι συντονισμένη και στην πραγματική τη ανθρωπιστική βοήθεια. Η σχέση μεταξύ του κατεπήγοντο και τη ανάπτυξη είναι εδώ πολύ έντονη, ιδίω σε μια χώρα όπου υπάρχει η ανθρωπιστική βοήθεια και δεν υπάρχουν οι κατάλληλε κρατικέ δομέ θα πρέπει ο πληθυσμό να έχει καλύτερη πρόσβαση στι βασικέ υπηρεσίε που οργανώνονται αυτή τη στιγμή από διεθνεί οργανώσει και μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τέλο, ε, η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν και στο update θα πρέπει να μα κάνει να ξεχνάμε την κατάσταση στον Ταρφούρο, που θεωρείται η μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια του, ε, κρίση γνώμη του κόσμου και θα ήθελα από την ευκαιρία να χαιρετήσω το έργο του κυρίου Μπάρς που μου φέρεται πάρα πολύ αξιόλογο. Ευχαριστώ κύριε Στρίφλα, λέει η πρόεδρος. Ο κύριος Χάουιτ, ένα μισή λεπτό. Θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να συνεργαστεί η Ένωση με τον Νότιο Σουδάν στον εκδημοκρατισμό. Θα είναι μια χώρα με όντως με εξαιρετικά υψηλό τον υψηλότερο δίκτυο παιδικής συνεισμότητας και τον χαμηλότερο ε, σχολικής εκπαίδευσης στον κόσμο. Γι' αυτό χρειάζεται παρέμβαση της Ένωσης. Η Ένωση λοιπόν θα έπρεπε να είναι περήφανη που συνέβαλε στην, ε, στο δημοψήφισμα και στην έκβασή του και πραγματικά να συγχαρώ και εγώ την κυρία Ντεκάιζερ για την δουλειά, την προσωπική δουλειά που έκανε. Έτσι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν Ένωση να βοηθήσουμε τον Νότιο Σουδάν και παραπέρα στην αναθεώρηση του συντάγματος, στην εφαρμογή πολυκομματισμού, στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η 9η Ιουλίου είναι η σημαντικότερη ημέρα για το Νότιο Σουδάν. Για το Βόρειο Σουδάν, ωστόσο, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις του σταματούν τότε. Πρέπει να μπορέσουν να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό και να αλλάξει η κατάσταση στο Νταρφούρ. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πίμπαρξ να μας εξηγήσει τι κάνει η Ένωση στη συνέχιση και επιδείνωση των ε, παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ε, ιδίως στην κράτηση ε, εκπροσώπων Σουδανών που ήταν ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Αποστολή. Εγώ είχα μετάσχει πρόεδρε στην ε, διαδικασία ανεξαρτητοποίησης του τιμό στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000. Ελπίζω η χώρα να προχωρήσει, το Νότιο Σουδάν να προχωρήσει με λιγότερα προβλήματα στην εξαρτησία, μια και έχει ήδη τραβήξει τόσα και τόσα. Ο κύριος Ρινάλντι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να συνοδεύσει κανείς τα πρώτα βήματα ενός νέου κράτους στα πλαίσια μιας ειρηνικής διαδικασίας. Θα πρέπει να διατηρήσει την ειρήνη αλλά να μην ε, ξεχάσει την ε, συνολική θα έλεγα αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο ΑΙΜΠΕΙ φαίνεται ότι υπονομεύουν τη θετική κατάληξη της διαδικασίας αυτής, αλλά αυτό θα δυσκολευτεί από την δημιουργία του 54ου Αφρικανικού κράτους στις αρχές Ιουλίου. Δεν θα πρέπει να χάσουμε από μπροστά μας την, τον βασικό στόχο που δεν είναι τόσο η ανεξαρτησία αλλά η δημιουργία αξιόπιστων θεσμών και η ανάπτυξη του πληθυσμού η οποία ζει βέβαια κατά 90% κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο πληθυσμός αυτός δεν την χάνει των μέχρι ακόμα αξένων ε, επενδύσεων ε, οι οποίες δεν θα είναι ληστρικές βέβαια όταν έρθουν ελπίζω και θα βοηθήσουν πραγματικά. Είναι ένα νέο μέτωπο λοιπόν το νέο Σουδάν, στα πλαίσια του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την αξιοπιστία που έχει πετύχει στην περιοχή. Ο κύριος Τάνοκ, ένα λεπτό. Στις 9 Ιουλίου θα, θα κηρύξει την ανεξαρτησία του, θα είναι ένα νέο κράτος, αγγλόφωνο μάλιστα. Οι επόμενοι μήνες λοιπόν θα είναι πάρα πολύ κρίσιμοι και το Νότιο Σουδάν θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ένα κυρίαρχο βιώσιμο κράτος αλλά ακόμα και χωρίς το βόρειο Σουδάν που είναι εχθρικό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν εχθρότητες διαφυλετικές, η υγεία είναι σε ικτρή κατάσταση, η εκπαίδευση αυτή, η οικονομία εξαρτάται πλήρως από την εξαγωγή πετρελαίου και γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε όλες τις μορφές βοήθειας προς τον Νότιο Σουδάν. Αλλά χρειάζεται και την πολιτική μας στήριξη τα προβλήματα που υπάρχουν στην συνοριακή περιοχή του Αμπιέ δείχνουν ότι ο πρόεδρος Μπασίρ δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει κοπεί στα δύο η χώρα του. Ελπίζω λοιπόν τα πράγματα να πάνε καλά στο Νότιο Σουδάν και θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα αναγνωρίσει ε, την ανεξαρτησία της Σομάλιλάντα. Ο κ. Σαγκουράκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε οι πρόσφατες συγκρούσεις στο αμπέι δείχνουν πόσο αβάσιμοι ήταν οι πανηγυρισμοί των ηπα και της ευρωπαϊκής ένωσης μετά το δημοψήφισμα. αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η υπεριαλιστική ειρήνη είναι εξίσου αιματηρή με τον υπεριαλιστικό πόλεμο. είναι προφανές ότι βορράς και νότος συντροχιά των υπεριαλιστών θύματα του ανταγωνισμού και της πολιτικής του διέρε και βασίλευε δύσκολα θα μπορέσουν να αποφύγουν μια ευθεία σύγκρουση το πετρέλαιο τα κοιτάσματα χρυσού χαλκού ουράνιου που διαθέτει το αμπιέι είναι αυτό που εδώ και 20 χρόνια επιχειρούν να εκμεταλλευτούν ποικίλε imperialistικέ δυνάμει. Αυτό ο ανταγωνισμό ευθύνεται για τον κίνδυνο ενό νέου ακόμα πιο αιματηρού πολέμου αφού τώρα θα υπάρχει άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω φαίνεται να επιδιώκουν οι ευρωενωσιακέ δυνάμει μετά και τον πόλεμο στη Λιβύη. Είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί τέρμα σε κάθε εμπεριαλιστική επέμβαση στο Σουδάν, σε κάθε πράξη εχθρότητα και αντιπαράθεση μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Εμεί πιστεύουμε ότι ο λαό του Σουδάν, στο Βορρά και στο Νότο, πρέπει να πάρει την τύχη στα χέρια του, μόνο έτσι μπορεί να αποφύγει τον πόλεμο και μόνο έτσι μπορεί να γίνει κυρίαρχο του πλούτου τη χώρα του για να προχωρήσει σε μια άλλη ανάπτυξη. Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ έχω την εντύπωση στου παρατηρητέ ε, του Κοινοβουλίου να είμαι παρόν στο δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν και πραγματικά με εντυπωσίασε η βούληση των Νότιων Σουδανών να ορίζουν ε, τη μοίρα τη χώρα του ε, στο μέλλον. Και πραγματικά μπορούσε να να ότι αισθάνονται ότι απελευθερώνονται από τη σκλαβιά. Ε, δεκάδες χιλιάδες εσωτερικά εντοπισμένοι άνθρωποι ξεκίνησαν να πάνε στη συμπαλιά τους νοτιοζωδανική πατρίδα. Θέλουν βέβαια σαν εξαρτησία της χώρας να ζουν σε ειρήνη και χωρίς διαμάχη με τους γειτονές τους όπου έχασαν εκατομμύρια τη ζωή τους στο παρελθόν. Σε νέα ηλίου θα είναι επίσημη η του Νότιου Σουδάν. Οι όροι κίνηση όμω είναι πάρα πολύ άσχημοι. Πολλά ελέγξαν πάνω σε αυτό. Το 70% ε, των, του πληθυσμού είναι ομάδε, το 80% είναι αναλφάβητοι. Η διαμάχη στο Αμπιχέ διευρύνει και γίνεται στρατιωτική. Διένυξε αυτή τη στιγμή με νεκρούς και τραυματίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν και ε, αντιπαλότητες μεταξύ διαφόρων φυλών στο νότιο Σουδάν και έχουν χάσει πολλοί ε, που έχασαν τη ζωή τους ε, από τον Γενάρη. Υπάρχει ο κίνδυνος η χώρα του Νοτιού Σουδάν να θεωρηθεί αποτυχημένη χώρα. Είμαι επιβεβαιωμένος ότι υπάρχει ευθύνη της Ευρώπης για την περιοχή αυτή λόγω του αφρικιακού παρελθόνου των χωρών αυτών. Μαζί με την ε, Αφρική Νοτιοαφρικανική Ένωση καλείται να δράσει η ευρωπαϊκή πολιτική όχι μόνο με χρήμα, αλλά και με την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών που αρχίζει να δημιουργείται εκεί. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να διαπραγματευτούν εκείνους που έχουν στα χέρια τους ε, την ε, μοίρα της χώρας αυτές, δηλαδή τους ε, φιλαρχούς και τις στρατιωτικές αρχές, για να μην απογοτεύσουμε τους πληθυσμούς. Ευχαριστώ κύριε Σέλερ. Η κυρία Κρετού, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ και πάνω από ένα, ε, σε λιγότερο από ένα μήνα θα γιορτάσει το Νότιο Ζωδάν την ανεξαρτησία του μετά από το δημοψήφισμα του Ιανουαρίου. Δυστυχώ το δημοψήφισμα αυτό δεν έλυσε τα προβλήματα όσον αφορά τα σύνορα και την κατανομή των πετρελαφόρων περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν να ενδυναμωθούν οι διπλωματικέ προσπάθειε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία του και η παρουσία των συναδέλφων, ιδίω τη κυρία Δεκάιζερ επιτόπου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κατάσταση έχει ε, επιδεινωθεί δραματικά. Πολλοί ε, αναγκάστηκαν να φύγουν από τις περιοχές στις ζούσαν και κινούμεθα προς μια ανθρωπιστική ε, κρίση. Χαίρομαι που αναφερθήκατε σε ρευτικές δυνάμεις στην περιοχή Υπάρχει και μια δήλωση της, ε, των Ηνωμένων Εθνών όπου αναφέρεται ακριβώς η αποτυχία της ε, στάσης των ε, στρατευμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Πριν λίγο καιρό, η κυβέρνηση του Σουδάν ενημέρωσε τον ΙΕ ότι οι προϋποθέσεις για την επιστροφή των αμάχων θα ξεκινούσαν. Από ό,τι γνωρίζουμε, γενικά ο κόσμος φεύγει γρήγορα αλλά γυρίζει με προβλήματα και κυρίως με σημαντικές ανθρωπιστικές και κοινωνικές ε, συνέπειες. Γι' αυτό προτείνω η Ένωση να θεσπίσει σύντομα μία αποστολή παρακολούθησης βάσει αυτό, αυτού που είχαμε κάνει στα Βαλκάνια με τη βοήθεια προφανώς της Αφρικανικής Ένωσης και ίσως και κάποιον τρίτων χωρών, γιατί όχι. Δύο λόγια τώρα για τις φήμες που ακούγονται για, την πιθανή, για μια πιθανή εθνοκάθαση στην περιοχή. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έπρεπε προφανώ να, να υπάρξει δράση της διεθνούς κοινότητας μετά από παρότενση της Ένωσης. Το δράμα της πρώην Ιουγκοσλαβίας δεν πρέπει να επαναληφθεί ουδόλως. Ο κύριος Πρέντα. Ένα λεπτό. Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και την δημιουργηθεί και τη δημιουργία του 54ου κράτους στην Αφρικανική Ήπειρο. Τώρα όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλάβουμε ότι η ειρηνική μεταξέλιξη του Σουδάν βρίσκεται σε κίνδυνο. 21 Μαΐου μπήκαν στην Αμπιγέη οι δυνάμεις του Σουδάν. Η βία αυξάνεται στο Καντουγκάλι χτες. Όλα αυτά δείχνουν ότι μπορεί να ξεκινήσει ο εμφύλιος μεταξύ Βορρά Νότου ανα πάσα στιγμή. Κάτι που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Πρέπει να είμαι σαφής. Οι άτακτες δυνάμεις και ο στρατός του Σουδάν ε, στο Αμπία και οι δύο, η παρουσία και των δύο, είναι παραβίαση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Ενισχύουν την βία. Η κατάσταση ασφάλειας πρέπει να λυθεί βάση της συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει κοινές, ε, την παρέμβαση δυνάμεων ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπάρχουν ερωτηματικά, συνεχίζουν να υπάρχουν ερωτηματικά για την ε, συνύπαρξη και των δύο κρατών. Χρειάζεται πολιτικός διάλογος. Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα κοινά σύνορα, ηθαγένεια, πετρελαϊκή πόρη. Πρέπει ταυτόχρονα να αποφύγουμε την επιδείνωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου. Ο Μαρ Μπασίρ συνεχίζει να είναι αντικείμενο ενός διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη οι αρχές. Μια θετική εξέλιξη είναι η απελευθέρωση των τριών Βουλγάρων ομήρων που δούλευαν για τον ΟΗΕ και που ε, ε απήχθησαν στον Ταρφούρ τον ε, Ιανουάριο. Μπαίνουμε στο Κάτς Ο κ. Μικολάσικ. Ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, ο εμφύλιος ο οποίος κράτησε για πάνω από 20 χρόνια στο Σουδάν, κατέστρεψε τη χώρα αυτή στο σύνολό της και σημάδεψε αρνητικά εκατομμύρια κατοίκων. Βέβαια ο πόλεμος αυτός ευτυχώς σταμάτησε τώρα, μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία είχε σαν προϋπόθεση το δημοψήφισμα. Η πρόληψη βέβαια είναι η καλύτερη μέθοδος και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει τα χρήματα που θα δώσουμε στο Σουδάν να μην ε, προορίζονται μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους ενός κράτους όπου οι κανόνες θα ισχύουν πραγματικά. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δείχνει ότι ο κυρίαρχα χριστιανικός νότος θέλει την ανεξαρτησία του. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γύρω από αυτό πια. Κυρία Νεβαλνόβα. Δεν Ανησυχώ για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή. Ιδιαίτερα η περιοχή του ΑΕΜΠΙΕ στην ουσία βρίσκεται σε 20 χρόνια πόλεμο η περιοχή αυτή. Από εκεί ξεκίνησε η σύγκρουση και μετά από τις δηλώσεις και της ε, Διεθνούς Ομάδας για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων οι εξελίξεις του IBF θα χαρακτηρίσουν το σύνολο των εξελίξεων. Θα οδηγηθούμε σε νέο πόλεμο, θα οδηγηθούμε στην ειρήνη. Πρέπει να στηρίξουμε την ειρήνη και γι' αυτό θα στηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταδικάζει τη χρήση βίας εις βάρος των πολιτών γιατί κάτι τέτοιο δυστυχώς οι πολιτοφυλακές εξακολουθούν να το κάνουν. Πολιτοφυλακές οι οποίες στην ουσία ήταν τα αφεντικά της περιοχής για πάρα πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να παίξει και πρέπει να το παίξει. Ζέμ και ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ένα σημαντικό πράγμα θέλω να πω. Όλοι εκφράζουμε τη χαρά μας, διότι ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος γεννήθηκε ένα καινούργιο κράτος, το Νότιο Σουδάν δηλαδή. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι μια ευκαιρία μόνο. Το κράτος αυτό σήμερα δεν έχει τα βασικά χαρακτηριστικά κράτους. Δεν έχει δομή, δεν έχει υπαλλήλου, δεν έχει δικαστές, Πολλοί δηλαδή μπορεί να εμπλακούν στην εξέλιξη υπονομεύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια. Πέραν της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να υπάρξει και καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας. Η κυρία Μπασέσκου. Ένα λεπτό. Καλωσορίζω την δήλωση της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής μετά τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Οι ηγέτες πρέπει να αποδεχθούν την, ε, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το Σουδάν έχει μακρά ιστορία βίας. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι υπάρχει μια επιστροφή στο παρελθόν. Θέλω να υπογραμμίσω την πολύ δύσκολη κατάσταση του πληθυσμού στις εμπόλεμες περιοχές. Είναι πιθανή μια ανθρωπιστική καταστροφή εάν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση. Επιπλέον, έγιναν επιθέσεις σε περιοχές που προστατεύονται από δυνάμεις του ΙΕ, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των στρατιωτικών και την επιστροφή των προσφύγων. Τονίζω την ανάγκη σταδιακού φοπλισμού των ομάδων που αρνούνται να δεχθούν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Οι εξελίξεις στην περιοχή υπονομεύουν την ε, διαδικασία εξαρτησίας. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Σκέλη, έχετε λόγο. Ναι, αυτή, το θέμα που συζητάμε σήμερα για το Σουδάν και τον Νότιο Σουδάν είναι ενθαρρυντικό και όλα αυτά έχουμε περισσότερα άσχημα νέα και όχι καλά νέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει μια νέα χώρα και να εξασφαλίσει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στο Σουδάν και κυρίως στο Νότιο Σουδάν. Ιδίως νομίζω ότι λόγω των ιδρυτικών ε, αρχών του Σούμαν που βασίζονται στην ειρήνη και στην ευμάρεια υπάρχει δυνατότητα ε, να μην έχουμε την εντύπωση ότι κάποιες χώρες εκμεταλλεύονται το Σουδάν για δικό τους σκοπούς εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης θα πρέπει να φροντίσουμε για τον νέο αυτό κράτο στο νότιο Σιδόν, δηλαδή κυρίω και να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν εμφύλιοι πόλεμοι όπως συμβαίνουν συχνά. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλωσίκο Βεμπένοβα. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μετά την ανεξαρτησία που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα έχει το του Σουδάν πολλά εσωτερικά ε, προβλήματα και οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό η εξωτερική βοήθεια στο νότιο Σουδάν ε, και το τέλος των ε, νόπλων συγκρούσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ήταν ήδη σημαντικό στο παρελθόν και παρόλο που πιστεύουμε ότι το νότιο Σουδάν θα ενταχθεί στη συμφωνία της Κοτονού Ε, θα υπήρχε ίσως εξ αυτού ένα κενό χρηματοδότησης και θα είναι πολύ ευάλωτο κράτος ε, το Νότιο Σουδάν και θα υπάρχει η περίπτωση, ή ο κίνδυνος κατάρρευσης του κράτους. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε τις Σουδανικές αρχές να ξεπεράσουν αυτή την δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ το στο λόγο κ. Μούσλε. Εκτός αυτή τη στιγμή υπάρχουν 50.000 ε, εκτοπισμένοι ε, και από την άλλη μεριά θέλουν ε, να γίνει στα γλίγορα ένα υποψήφιο στο ABA με την υποστήριξη του στρατού. Πολύ περίεργες καταστάσεις δηλαδή. Δεν είναι θέμα μόνο διαφορετικές αντιμετωπίσεις του ιδιοκτησίας που οδηγούν στα προβλήματα αυτά του ABA. Υπάρχουν και διαφορετικές ε, θρησκείες γιατί υπάρχει ο Βορράς που είναι μουσουλμανικός και ο Νότος είναι χριστιανικός και είχαν ενωθεί λόγω των απεικονατικών ε, συνόρων. Δεν θα έπρεπε να είχε γίνει στα γλίγορα τόσο πολύ γρήγορα το δημοψήφισμα εφόσον ήταν γνωστό τι θα γινόταν με τους ε, ψηφοφόρους του ΑΜΠΙΕΙ. Έχουν παρευρεθεί πολλές περιοχές και αυτό δεν επιτρέπεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μέσλερ. Τελευταίο είναι ο κύριο Ζάλερ. Ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ δεν είχα ποτέ εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Πασίρ και ούτε του έχω και τώρα. Είμαι απεσιόδοξος ότι το Σουδάν δεν θα επαναλάβει τα σπάνωτα του παρελθόντος και δεν ξέρω τι θα γίνει, κατά πώς θα υπάρχει παρέμβαση στο Νότιο Σουδάν ή θα προσπαθήσει να καταλάβει κάποιους πόρους πλούτου, τι έχει προετοιμάσει δηλαδή προληπτικά η Κομισιόν για το θέμα αυτό σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και την ε, Νοτιοαφρικανική Ένωση. Και επίσης ήθελα να ξέρω ποια είναι τα τμήματα που θέλετε να αναλάβετε εάν κάτι τέτοιο συμβεί. Αν δηλαδή το Βόρειο Σουδάν καταπατήσει την συνθήκη ειρήνης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριο Σπάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. το Σουδάν είναι μια χώρα που ψήφιζε να γίνει ανεξάρτητο, το Νότιο Σουδάν δηλαδή. Το τελευταίο κράτος, το πιο πρόσφατο μέλος το ΙΕ θα γίνει. Εξαρτάται πολύ σωστόσο από τον βόρειο γείτονά του, αλλά και από την Ένωση και τα άλλα αφρικανικά κράτη. Στο κράτος αυτό ο κόσμος δεν περιμένει να δεν είναι συνηθισμένο στο να δουλεύει, αλλά στο να πολεμάει. Οι μόνοι που δουλεύουν είναι οι γυναίκες και τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο. Γι' αυτό και το Νότιο Σουδάν δεν έχει δάσκαλους, δεν έχει γιατρούς. Πρέπει να χτιστεί το κράτος από τα θεμέλια, να αποκτήσει λειτουργικό πολιτικό σύστημα, να υπάρξει Κύριε Πίτρο, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας, για τη στρατηγική την οποία ακολουθήσατε. Λίγα στοιχεία θα ήθελα να σχολιάσω από αυτά που υπόθηκαν. Οι ηγέτες της περιοχής είναι οι λαοί του Νοτίου και του Βορείου Σουδάν. Εμείς ε, ε, βοηθούμε τις διαδικασίες που επιλέγουν. Βέβαια δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση σήμερα μετά το δημοψήφισμα. Υπάρχει βία, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είναι διαφορετικού επίπεδου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε φως στον άκρη του τούνελ. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μας για μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, γιατί υποστηρίξαμε τη διαδικασία αυτή και πολιτικά και με τις δράσεις μας και με την οικονομική μας παρέμβαση. Εμείς ποτέ δεν υποχωρήσαμε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο θέμα του διεθνούς ποινικού. Εμείς έχουμε ξεκάσαρες θέσεις και για τα δύο αυτά θέματα. Όποτε υπάρχει παραβίαση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ύπατη εκπρόσωπος για τα εξωτερικά θέματα κάνει άμεσες παρεμβάσεις. Θα μου πείτε ότι δεν υπάρχουν άμεσες ε, αντιδράσεις από την περιοχή. Παρ' όλα αυτά επιμένουμε. Για το ΆΜΠΙ η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη καταδίκη της ε, κατάστασης εκεί και να ζητήσουμε ε, άμεσα να επιληθεί το πρόβλημα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ένας χώρος στον οποίο θα αποφασιστεί αν θα υπάρξει μια νέα αποστολή. Και αν ναι υπάρξει μια τέτοια απόφαση, ένα τέτοιο ψήφισμα, θα την υποστηρίξουμε. Θεωρούμε όμως ότι η ισχυρή, ισχυρή συγγνώμη, πολιτική μας θέση είναι αυτή την οποία σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να διαφορφώσουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα που έδωσα στο Νότιο Σουδάν. Μην πιστεύετε ότι όλα αυτά τα θέματα θα επιληθούν στις 9 Ιουλίου. Σίγουρα θα ανακηρυχθεί ανεξαρτησία, αλλά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και αυτό που έχει σημασία είναι το πάνελ της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης να υποστηριχθεί και από τις δύο πλευρές, και από το Βορρά και από το Νότο και εμείς θα υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι τα δύσκολα θέματα θα τύχουν απαντήσεων. Τώρα για το θέμα του χρέους. Υπάρχει προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τις φτωχές χώρες και υπάρχει άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση. Δεν το έχουμε ξεχάσει το θέμα. Για το θέμα της Κίνας. Κοιτάξτε, όσο μπορούμε να εμπλέξουμε την Κίνα, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και καλό θα είναι να βρούμε λύσεις και με τη βοήθειά της, αλλά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Έχουν υπάρξει δραστηριότητες ε, των Κινέζων στην περιοχή, σε ορυχία, στο πετρέλαιο και η διεθνής κοινότητα με την Κίνα θα πρέπει να βρει λύσεις. Τέλος, σας είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον σας για το Σουδάν. Το Σουδάν είναι μακριά μας βέβαια, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι τόσο μακριά. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και ο κόσμος συνεχίσει να πεθαίνει στην Αφρική, η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει ότι δεν ξέρει και να λέει ότι είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρύνετε και την κυρία Άστον και εμένα έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι προσπάθεια ε, γίνεται για να ε, ζήσει ο λαός της περιοχής εν ειρήνη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κλείνουμε τώρα τη συζήτηση. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί, θα ψηφιστούν στις 12 την Πέμπτη. Προχωρούμε τώρα στην εξέταση της έκθεσης